Ε, συνεδρίαση ε, τη 11 η Νοεμβρίου είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι. Κατόπιν τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά.